Στο στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση τη ΥΠΑ εκπροσώπου της για εξωτερικέ υποθέσει και πολιτική ασφαλεία, την Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναφερθεί στην κατάσταση στο Ιράκ. Σα ξαναδίνω λοιπόν το λόγο Βαρόνι Άστον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άμα δούμε το Ιράκ σήμερα, Βλέπουμε πραγματική πρόοδο, παρά το γεγονό ότι είναι πολλαπλέ οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή. Θέλω να εστιάσω όμω την παρέμβασή μου στο μέλλον του Ιράκ σε μια χώρα με μεγάλη δυναμικότητα και πολλά που έχει επιτύχει στο παρελθόν. Η βία στο χαμηλότερο επίπεδο τη από το 2003, παρά το γεγονός ότι είδαμε πολύ σημαντικές επιθέσεις κατά κυβερνητικών κτηρίων, ο αριθμό των θυμάτων των αμάχων το 2009 ήταν λιγότερο από το μισό των θανάτων το 2008. Η διαφατριακή βία ήταν πολύ μικρότερη από τις εποχές του 2006-2007. Το Ιράκ έχει ένα νέο σύνταγμα και έχει <clears throat> προχωρήσει σε εκλογές με σημαντική συμμετοχή του πληθυσμού παρά τους κίνδυνους. Χάρη στο θάρρος του λαού του Ιράκ, οι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν ριζώσει εκεί. Οι περιφερειακές εκλογές πέρσι λειτουργήσαν πολύ ομαλά σε όλο το Ιράκ οι επόμενες γενικές εκλογές που θα γίνουν σε 7 Μαρτίου 2010 μπορούν να αποτελέσουν ένα περαιτέρω ορόσημο για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε τη δημοκρατία στο Ιράκ. Από τη δική μας πλευρά αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειε μα υποστήριξη του Ιράκ θα πρέπει να συνεχιστούν και θα πρέπει να επεκταθούν και σε νέε περιοχέ όσο βελτιώνεται η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ βοήθεια προ το Ιράκ από το 2003 μέχρι σήμερα για την υποστήριξη βασικών υπηρεσιών, ανθρώπινης ανάπτυξης, προσφύγων, ευκυβερνησίας και δημιουργίας ικανοτήτων. <clears throat> Όλα επί τη βάση των προτεραιοτήτων του ίδιου του Ιράκ. Η ολοκληρωμένη μας αποστολή για το κάτω δικαίου, η U-Just, έχει παραταθεί πολλές φορές αιτήσει του Ιράκ και τώρα εκπαιδεύει και άτομα μέσα στο Ιράκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των εκλογικών διαδικασιών. Θα συνεχίσουμε και στο Ιράκ και σε άλλε περιοχέ μέχρι ότου οι αρχέ του Ιράκ μπορούν να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη αυτών των διαδικασιών. Υπάρχει μια σημαντική πρόοδο και γι' αυτό εμεί δίνουμε όλο μεγαλύτερη ε, σημασία στο να συμμετέχουν οι Ιρακινοί και να υπάρξει βιωσιμότητα αυτή τη ε, διαδικασία. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόηση για την ενεργειακή συνεργασία και θα υπογράψουμε συντόμω μια συμφωνία συνεργασίας. Είναι η πρώτη συμβατική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ. Θα καλύψει θέματα από πολιτικό διάλογο μέχρι το εμπόριο, ρυθμιστική, συνεργασία ρυθμιστικών αρχών και αναπτυξιακή βοήθεια. Θέλουμε μια βαθύ, ένα βαθύτερο και ευρύτερο πολιτικό διάλογο με το Ιράκ που θα καλύπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ιρακινό Κοινοβούλιο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιράκ και περιμένουμε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Εκπροσώπων του Ιράκ στο μέλλον. Το Ιράκ θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις πολλαπλές προκλήσεις. Οι εκλογές της 7ης Μαρτίου θα είναι σημαντικές, θα πρέπει να είναι αμερόληπτες και ελεύθερες. Εμείς θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία. Θα στείλουμε μια ομάδα αξιολόγηση των εκλογών στο Ιράκ για να αναλύσει την εκλογική διαδικασία και να προβεί σε συστάσεις και προτάσεις το Ιράκ βρίσκεται σε θετική τροχιά, είμαι σίγουρη θα χρησιμοποιήσει τους νέους θεσμούς του για να βρει τις απαραίτητες συμβαστικές λύσεις που θα οδηγήσουν στην εθνική συμφιλίωση. Από τη δική μας πλευρά, εμεί θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε το Ιράκ και θα το υποστηρίξουμε μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Προσβλέπω λοιπόν στην συζήτηση που θα λάβει η χώρα. Σα ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση με τους αγορητές που εκπροσωπούν τις ομάδες τους. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ντελάγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ύπατη εκπρόσωπο για τα λόγια που μας απίφθινε. Ε, αντίχησαν ε, αισιόδοξα, θετικά τα μηνύματα. Εσείς ε, επισημάνατε τον χαμηλότερο αριθμό των νεκρών αλλά ακόμα και οι ανώθευτες εκλογές ε, δεν ε, ταυτίζονται με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η πλειοψηφία δεν σημαίνει ότι είναι πλέον ε, σαφές ε, ποιος έχει δίκιο. Μια όρημη δημοκρατία αναγνωρίζει και τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι στη δήλωσή σας δεν άκουσα τίποτα για τις ε, μειοψηφίες. Γιατί ανησυχώ. Η Human Rights Watch λέει ότι διώκονται ακόμα οι μειονότητες. Από το 2005 είχαμε 65 επιθέσεις σε χριστιανικές εκκλησίες ο πατέρας ε, δύο κοριτσιών δολοφονήθηκε στο δρόμο καθότι ήταν χριστιανός. Πολλοί χριστιανοί εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το Ιράκ. 500.000 μετά την εισβολή των ε, Αμερικανών και 350.000 εξ αυτών ε, μάλλον 100.000 έχουν παραμείνει πρόσφυγες. Στο άρθρο 2 της συνθήκης ε, γίνεται λόγος για τα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και αυτά θεωρούνται ε, θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Χρίζουν του σεβασμού μας. Εσείς λοιπόν κυρία Άστον πρέπει να διεκδικήσετε αυτό το σεβασμό σε διεθνές επίπεδο. Μέχρι τώρα η Κομισιόν εξαρτάτο από τη διεθνή βοήθεια από τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Εσείς ε, λέτε ότι υπάρχουν προτεραιότητες για το Ιράκ. Θα ήθελα όμως να ακούσω από εσάς την ίδια πώς σκοπεύετε να μεριμνήσετε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει καλύτερα όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια στο Ιράκ. Και θα ήθελα να ακούσω παρακαλώ την άποψή σας επ' αυτόν. Σας ευχαριστώ για την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Για δύο λεπτά, κυρία Κώστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Άστον, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει αυτή τη συζήτηση ενώπιση των εκλογών του Μαρτίου στο Ιράκ. Η διαδικασία πολιτική στο Ιράκ θα δείξει, όπως, εάν όπω λέγατε εσεί, ε, θα δούμε κατα... ότι είναι εύθραυστη η διαδικασία, οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε τους νέους θεσμούς της χώρας και την πολιτική ισορροπία στην οποία βασίζονται. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαν στόχο, αν θέλουμε να φτάσουμε στην πρώτη απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων τον Αύγουστο, διότι χωρίς αυτό, θα, τα θέματα υπήρχαν προβλήματα. Οι σύγκρουση μεταξύ Σουνιτών, Σιητών και ε, Κούρδων πρέπει να διευθυνθεί, θα χρειάζονται νέοι νόμοι για να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα. Τώρα, ε, δημιουργούνται ανησυχίες και θα θέλαμε την άποψή σα για την πρόσφατη απόφαση τη Εκλογική Επιτροπή. Πολλοί υποψήφοι και κόμματα να μείνουν εκτό. Αυτοί που είναι πιο κοντά στου Σουνίτε ή στου Χριστιανού, ούτω ώστε μπορεί να αποδυναμωθεί η δημοκρατική διαδικασία στο Ιράκ, που είναι αδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των δράσεων που έχουν αναλυφθεί. Θα πρέπει να ακολουθήσει, παρακολουθήσει την, την εκλογική διαδικασία όπω υπόθηκε, αλλά να βρέχει πιο σημαντικέ φιλοδοξίε. Θα πρέπει ε, το κοινοτικό πρόγραμμα Eurojust Lex ε, μπορούμε να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις θεσμούς, ε, δημοκρατικούς θεσμούς στο Ιράκ και την νομοθεσία στο Ιράκ και σαν ομάδα πιστεύουμε ότι είναι θετικό το ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την διάρκεια της αποστολής ε, μέχρι 30 Αυγούστου του 2010. Πρέπει να δώσουμε υποστήριξη στο Ιράκ μέσω του προγράμματος συνεργασίας με στόχο τη συμμετοχή στη διαδικασία σταθεροποίησεως ε, της χώρας ενισχύοντα μετά από τις ε, εκλογές, τις επαφέ μεταξύ των κοινοβουλίων. Πολλά κράτη-μέλη συνεργάζονται με το, ε, με το Ιράκ. Έχει σημαντικό πρόγραμμα πολιτιστικής συνεργασίας Ιταλία από το Ιράκ. Λοιπόν, η πολιτική ισορροπία στο Ιράκ είναι σε σημασία όχι μόνο για τη χώρα αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει στρατηγικά στην περιοχή το Ιράκ για να ξεπεραστούν υπάρχουσε συγκρούσει και να εξασφαλιστεί με δηλωθεί η ειρήνη. Γι' αυτό η βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία από πλευρά τη περιφερειακή κυβερνήσεω του Κουρδιστάν είναι ένα θετικό βήμα προόδου προ αυτή την κατεύθυνση. Ράκ παραμένει, όπω γνωρίζουμε, μια χώρα με σοβαρότερα προβλήματα ασφαλεία όσον αφορά τη σεβασμό δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχει και ανασφάλεια οικονομική. Υπάρχουν ε, οι πρόσφυγε, το 10% του πληθυσμού που είναι ευάλωτε ομάδε. Υπάρχουν εθνοτικέ ομάδε, οι γυναίκε, οι διάφορε εθνικέ μειονότητε και τα παιδιά, όλα αυτά υπόκειται σε αρνητικέ συνέπειε καταστάσεω. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ακόμα να έχουμε καλύτερο ρόλο ε, μέσω υποστηρίξεω προς μη κυβερνητικές οργανώσεις και ευρωπαϊκές οργανώσεις και ντόπιε και οι γυναίκε θα μπορούσαν στρατηγικοί φορεί για να ξεπεραστούν ε, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για Βαντάλεν, για δύο λεπτά, ε, για την πολιτική του ομάδα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιπάτη, εκπρόσωπος, είναι γεγονό ότι το Ιράκ δεν είναι εξασφαλισμένο, δεν είναι ασφαλές. Αν δούμε το Ιράν, το Ιράν προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του περισσότερο από ό,τι απαιτείται στο Ιράκ. Σε όλο το νότιο τμήμα του Ιράκ με την υποστήριξη της ηθικής μειονότητας. Δεν άκουσα την Υπάτη να ομιλά για το Ιράν, την Ιπάτη εκπρόσωπο εννοώ. Πώς βλέπετε λοιπόν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιορίσει την επιρροή του Ιράν και να μην το αφήσει να επεκταθεί στο Ιράκ. Αν μιλάμε για το βορρά του Ιράκ, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ της Τουρκίας και το Ιράκ σε σχέση με την περιοχή του Κουρδιστάν. Φυσικά, μπορεί να υπάρξει νομιμότητα στις προσπάθειες της Τουρκίας να αντιμετωπίσει τους αντάρτες οι οποίοι απειλούν την Τουρκία, αλλά εκεί περιορίζεται η δυνατότητα δράσης της Τουρκίας. Η αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ πρέπει να έχει την αυτόνομη της ανάπτυξη. Αν μιλήσετε για το ενεργειακό μνημόνιο κατανόησης, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το Ιράκ δεν είναι ένα ενιαίο κράτος. Το μνημόνιο αυτό θα πρέπει να συζητηθεί επίσης και με την αυτόνομη κυβέρνηση του κουρδικού τμήματος, γιατί υπάρχει ακόμα το θέμα του ποιος θα πρέπει να έχει την κατοχή των πετρελοπηγών της Κυρκούκ. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ δεν είναι ακόμα σωστά εκπαιδευμένες και δεν λειτουργούν σωστά. Δεν πρέπει λοιπόν μονάχα να υποστηρίξουμε το κράτος του δικαίου, αλλά εάν είναι απαραίτητο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε για να εξασφαλίσουν την <clears throat> ασφάλεια στο Ιράκ. Αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ενέργεια, οικονομία, σταθερότητα, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τα κράτη που είναι όμορα του Ιράκ. Παρακαλώ λοιπόν να έχετε μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. Για δυόμιση λεπτά δίνουμε το λόγο στην κυρία Evans, εκ ομάδας της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστήσω την ύπατη εκπρόσωπο, την Βαρόνη Άστον για τις δηλώσεις τη. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τη συζήτηση που δεξάγεται απόψε λαμβάνει η χώρα έναντι του ιστορικού της έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον παράνομο πόλεμο στο Ιράκ. Τι μπορούμε να μάθουμε από εκεί και πολλές πληροφορίε έρχονται στο φως που επιβεβαιώνουν αυτά που πιστεύαμε πολύ τότε που έγινε η εισβολή, ότι ο λόγος για τον πόλεμο ήταν το αλλαγή καθεστώ και έλεγχο των πόρων και όχι απειλή ε, υπάρξεω όπλων μαζική καταστροφή. Και όσον αφορά μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το μεταπολεμικό Ιράκ, οι λέξει όπω ε, πολύ άσχημα, ε, πολύ ανεπαρκή μέτρα χρησιμοποίησαν όλοι οι αρμόδιοι όσον αφορά την κατάσταση. Βλέπουμε τώρα σοβαρέ συνέπειε τη δράση. Η Βαρόνια Άστον είπε ότι κάποια πρόοδο έχει επιτευχθεί και βεβαίω επετέχθη, αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που απομένουν. Δεν υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των μειονοτήτων στο Ιράκ. Συνεχώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα προσφύγων. Οι συνδικαλιστέ, δημοσιογράφοι, γυναίκε πολιτικοί και οι υπασπιστέ με συγχωρείτε, διακόπτη πρόεδρο, μπορεί να μιλάτε πιο σιγά, διαφορετικά Διαρμηνεί δεν καταφέρω να σα ακολουθήσω πιο σιγά, πιο αργά. Αλλιώ οι διερμηνείς δεν μπορούν να σα ακολουθήσουν. So well, sorry. Trade union. Οι συνδικαλιστέ, οι δημοσιογράφοι, οι γυναίκε, πολιτικοί και οι υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαφανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν. Επιθέσει αυτοκτονία συνεχίζονται. Με τι εκλογέ που θα γίνουν στι 7 Μαρτίου, η Επιτροπή Εκλογών του Ιράκ την περασμένη εβδομάδα απαγόρευσε περίπου 500 υποψηφίου κυρίω πολιτικού Σουνίτε, που δεν συμμετάσχουν ήδη υποεκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο του Ιράκ και αυτό σίγουρα θα οδηγεί σε μεγαλύτερες εντάσεις και αστάθεια. Και τον περασμένο Νοέμβριο η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παρότρινε την κυβέρνηση του Ιράκ να αναστείλει τη θανατική ποινή και να την καταργήσει. Αλλά 900 άνθρωποι περιμένουν ακόμα να εκτελεστούν στο Ιράκ και πολύ συχνά ε, λαμβάνονται ε, θανατικές, ε, αποφάσει για θανατικές ποινές, μια πρόσφατα ελήφθη μάλιστα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε οικοδόμηση δημοκρατίας και να γίνονται σεβαστά ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Και ε, πρέπει να έχουμε τι προτεραιότητε στι συνομιλίε με το Ιράκ. Θα πρέπει να υπάρχουν βασικέ επίση παρέχοντε, όπω είναι η παιδεία και η υγειονομική περίθαλψη. Το κράτο δικαίου πρέπει να κρατήσει και θα πρέπει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να υποστηριχθεί. Η συνεργασία, η συμφωνία Συνεργασίε και τελική σχέση θα πρέπει να είναι βάση και μελλοντικέ εργασίε. Θα πρέπει να ζητήσουμε άμεση δράση σε θέματα όπω είναι η κατάργηση τη θανατική ποινή όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων ομάδων που είναι στόχοι και ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ για τους συντηρητικού και ευρωπαίους μεταρρυθμιστές. Το λόγο έχει ο κύριος Στίβενσον για ένα λεπτό. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, Βαρόνι Άστον, οι εκλογές ε, δεν θα είναι ελεύθερες και αδιάβλητες ε, στο Ιράκ. Πριν από δέκα μέρες αποφασίστηκε να απαγορευτεί ο επικεφαλής ενός κόμματος που ήταν και μέλο στο Κοινοβουλίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το απαγορεύτηκε λοιπόν να συμμετάσχει στις επικείμενες εκλογές και δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι αυτή η εξοργιστική απαγόρευση συνέπεσε και με την απαγόρευση πάρα πολλών άλλων πολιτικών στο Ιράκ την ίδια μέρα όπου ε, ο Πρωθυπουργός επισκεφτόταν την, ε, Πρωθυπουργός Σαντάν επισκεφτόταν την Βαγδάτη. Οι μουλάδες ε, επιμένουν τώρα στο να απαγορευθεί σε κάποιους πολιτικούς στο Ιράκ να συμμετάσχουν. Ο κύριος Μπάιντεν βέβαια έχει ήδη διαμαρτυρηθεί και ελπίζω κυρία αστόν ότι θα το πράξετε και εσείς αυτό γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα έχουμε πάλι ένα κράτος μουλάδων και με το τον τρόπο αυτό δεν θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την νομιμοποίηση των εκλογών. Σας ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την κυρία Άστον. Επιτρέψτε μου να μην συμμερίζομαι βέβαια την αισιοδοξία σας Καλό είναι ένα είναι αισιόδοξο κανεί στη ζωή, αλλά με το Ιράκ και με την κατάσταση που έχουμε δεν χωρεί περιθώριο για αισιοδοξία. Η απόδειξη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην στείλει παρατηρητές γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφαλειά τους. Αυτό είναι εύγλωτο. Αυτό δείχνει ποια είναι η κατάσταση με το Ιράκ. Δεν θέλετε να μιλήσετε για το παρελθόν, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε μια χώρα η οποία έχει εξανδραποδιστεί με ένα εκατομμύριο νεκρούς, τέσσερα εκατομμύρια εκτοπισμένους, μια χώρα που έχει ένα άδικο καθεστώς το οποίο βασίζεται σε ψέματα. Δεν υπήρχε ούτε σύνδεση του Σαντάμ Χουσέ με την Αλκάιντα, ούτε όπλα μαζική, μαζικής καταστροφής. Το μόνο που υπήρχε ήταν το συμφέρον των Αμερικανικών εταιριών να βάλουν χέρι στο πετρέλαιο του Ιράκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί λοιπόν <clears throat> να συνεχιστεί κάτω από τις δυνάμεις κατοχής. Η παρουσία του στρεβλώνει τα πάντα. Δεν με εκπλήσει ότι η απόφαση που ελήφθη να απαγορευτούν κοσμικά κόμματα μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική εσωτερική αντιπαράθεση. Υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές πρεσβείες οι οποίες δεν αποκλίνουν και τη δυνατότητα ενός στρατιωτικού πραξικοποιήματος μέσα στο Ιράκ. Είναι πάρα πολύ αρνητική κατάσταση. Εγώ θα σας ζητήσω να εργαστείτε με ταχύτητα ώστε το ταχύτητο δυνατό να φύγουν οι δυνάμεις κατοχής γιατί η παρουσία τους στρεβλώνει τα πάντα στο Ιράκ. Θα πρέπει λοιπόν οι Ηνωμένες, τα Ηνωμένα Έθνη να εξασφαλίσουν την επαναφορά στην ομαλότητα και να σταματήσει κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Για την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, ο κύριος Μπέλτερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον. Τα Χριστούγεννα του 2009 πολλές εκκλησίες στο Ιράκ έκλεισαν γιατί υπήρχαν απειλές ε, για τοποθέτηση βόμβας και αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη χρονιά και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Πολλές εκκλησίες ε, παραμένουν άδειες γιατί όλο και περισσότεροι χριστιανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η βία που της βάρος τους είναι όλο και πιο έντονη. Ε, πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε τρεις ε, θανατηφόρες επιθέσεις στο Κυρκούκ όπου παλαιότερα οι χριστιανοί ήταν ασφαλείς. Τώρα υπάρχουν όλο και περισσότερες απαγωγές και δολοφονίες και γι' αυτό πολλές οικογένειες οικογένειες χριστιανών ε, φεύγουν, εγκαταλείπουν τη χώρα. Ε, πριν από κάποια χρόνια στο Ιράκ Είχαμε περίπου 3 εκατομμύρια χριστιανούς. Ε, τώρα δυστυχώς μετά από καθαρίσεις θρησκευτικής φύσεως που έλαβαν χώρα οι άνθρωποι αυτοί αμαγκάστηκαν να φύγουν η αφγανοποίηση του Ιράκ δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Εσείς τι έχετε να πείτε από αυτού, ε, κυρία Άστον. Είναι μια χώρα όπου αν δεν υπάρχει εκεί η ε, χριστιανική κοινωνία δεν θα υπάρχει και ανεκτικότηση και αυτό θα είναι σίγουρα επιζήμιο για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ξεκινούμε το κατάλληλο με τα ονόματα των άλλων αγοριτών. Σας παρακαλώ όμως να σεβαστείτε το χρόνο στη διάθεσή σας, διότι έχουμε κάποια καθυστέρηση. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Μπαντέσκου. Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, κυρία Πρόεδρε, οι εκλογές της 7ης Μαρτίου έχουν οδηγήσει σε μια συμμαχία πολιτικών δυνάμεων στο Ιράκ. Ορισμένοι θέλουν να υπάρξει ένας ευρύτερο συνασπισμό στο Ιράκ. Ο Πρωθυπουργό του Ιράκ προσπάθησε να φέρει ανεξάρτητους υποψηφίους στο συνασπισμό αυτό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μετά από τις εκλογές αυτές θα πρέπει να οργανωθεί και ένα δημοψήφισμα για το καθεστώς της Κερκούκ. Είναι γεγονό ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στο Ιράκ. Έχουν διαμφισβητήσει πάρα πολύ και την διαδικασία την εκλογική στο Ιράκ και έχουν δημιουργηθεί εντάσεις. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται η Βαγδάτη είναι το εξή. Το δημοψήφισμα για τη σχέση με, την, ε, με με τις Ηνωμένες Πολιτείες η ρύθμιση των θεμάτων των, των ε, πετρελαϊκών πόρων, το γεγονός ότι υπάρχουν 900 άτομα επί των οποίων επικρέμαται η θανατική ποινή, οι βασανισμοί, η επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξάλλου η, το υψηλό επίπεδο διαφθοράς. Παραδείγματο χάρη, η σύλληψη του προηγουμένου Υπουργού Εμπορίου, του πρώην Υπουργού Εμπορίου στο Ιράκ. Η Ρουμανία προσπαθεί να βοηθήσει αυτήν την μετάβαση από το στρατιωτική κατοχή στην ε, πολιτική διακυβέρνηση. Χρειάζεται όμως και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γκόμες έχει το λόγο για μισή λεπτό. Όσοι έχουν οι καταστάσεις ασφαλείας στο Ιράκ δεν έχουν καταφέρει να εδρεωθούν οι δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού του Ιράκ. Υπήρξε πρόσφατα μια προσπάθεια δημιουργίας ευρύτερης συμμαχίας και συνασπισμού στο Ιράκ για να υπάρξει μια λύση των προβλημάτων τη χώρα αυτή. Το γεγονό ότι υπάρχει ένα νέο κουρδικό κόμμα δείχνει ότι υπάρχει μια ομαλοποίηση τη κατάσταση στο Ιράκ. Αλλά αν υπάρξει επιβεβαίωση ότι πάνω από 500 Σουνίτε πολιτικοί έχουν αποκλειστεί από τι εκλογέ, αυτό δεν θα βοηθήσει την συμφιλίωση σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση των εκλογών και εσωτερικέ αντιπαραθέσει. Επίσης το θέμα της θανατικής ποινής. Οι Ευρωπαίοι, κύριε θα πρέπει να πείσουν τις αρχές του Ιράκ να καταργήσουν την θανατική ποινή και είναι σημαντικός και ο ρόλος της ULEX εκεί. Υπάρχει ακόμα πάνω από ένα εκατομμύριο Ιρακινών που βρίσκονται σε όμορες χώρες. Κάποιοι από αυτούς δεν θα μπορέσουν ποτέ να γυρίσουν στο Ιράκ. Τα κράτη που έκαναν την εισβολή στο Ιράκ το 2003 έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για όλους αυτούς τους πρόσφυγες για την, τα θέματα των ανθρώπων αυτών, όπως και της υποστήριξης των ΜΚΙΟ, των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της διαφθοράς, θα πρέπει να επιτρέψει η Ιρακινή κυβέρνηση την ελεύθερη οργάνωση της κοινωνίας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ελεύθερη επαφή μεταξύ των Ιρακινών ΜΚΙΟ και των Ευρωπαϊκών. Είναι απαραίτητη μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών για να μπορέσει να δρεωθεί η δημοκρατία στο Ιράκ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για ένα λεπτό ο κύριος Πορέμα. Σας παρακαλώ, διαβάζετε πιο αργά τις παρεμβάσεις. Διαφορετικά, οι διερμηνείς δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, Βαρόνι Άστον. Το θέμα που συζητάμε μας δείχνει ποια είναι η κατάσταση. Γίνονται διεθνεί προσπάθειες στο Ιράκ. Αν δείτε και τι αραβικές προσπάθειες που καταβάλλονται, γίνονται προσπάθειε γενικά. Αλλά γίνονται επιθέσει ακόμα, πιέζεται η θρησκευτική μειονότητα και άλλες θρησκευτικέ μειονότητε. Και δεν νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όλα τα μέτωπα πρόσφατα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις αποσταθεροποιούν το Ιράκ και αυτό έχει αντίκτυπο ευρύτερο σε όλη την περιοχή. Μπορούμε να κερδίσουμε πολλά από μια αποκατάσταση της σταθερότητας στο Ιράκ και βεβαίως υπάρχει και η Ιρανική διάσταση στο θέμα. Νομίζω ότι τίθεται ένα θέμα όσον αφορά τις προσπάθειες του Ιράν να επηρεάζει τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει ο τρόπος στο Ιράκ. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Να ασκήσουμε πιέσεις. Να σταματήσουμε το Ιράν από το να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στις υποθέσεις του Ιράκ. Και αυτό θα ανοίξει την πόρτα σε σχετική σταθεροποίηση της χώρας, πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, επόμενος ο μιλητής, ο κ. Μελασσόν. Κυρία... Κυρία Υπάτη, εκπρόσωπος, η αισιοδοξία σας σε ό,τι αφορά την κατάσταση του Ιράκ και στην ε, κυβερνούσα πλειοψηφία δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Το Ιράκ έτυχε εισβολής μετά από μια ψευδή ε, φημολογία σε σχέση με όπλα μαζικής καταστροφής. Έχει λαιλατηθεί η χώρα αυτή, έχει διχαστεί ο πληθυσμός, υπάρχει θρησκευτικός φανατισμός που οδηγεί σε περισσότερους ριζοσπαστικούς αγωνιστές. Η κατάσταση είναι απόλυτα ικτρή και άδικη. Τι θα κάνετε για να ζητήσετε λογαριασμούς στους υπόλογους της χώρας οι οποίες ευσέφθησαν και οι οποίες είναι έτοιμες αύριο να το ξανακάνουν στην Ιεμένη ή κάπου αλλού ποια μέτρα θα λάβετε για να καταδικάσετε την χρήση σε ε, χημικών και βιολογικών όπλων και απεμπλουτισμένου ουρανίου που καταστρέφουν την υγεία όλων των γενναίων στο Ιράκ. Γιατί νομίζετε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα και στο Αφγανιστάν όταν δεν κοιτάζουμε το Ιράκ. για ένα λεπτό. Προβέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε με τις ε, εκλογέ, χαιρόμαστε να γίνουν εκλογέ ε, προσεχώ στο Ιράκ, διότι είναι άλλο ένα βήμα προ τη δημοκρατία. Δεν θα είναι ελεύθερε και δίκε, αλλά θα πρέπει να αρκεστούμε ε, για ένα μικρό βήμα που γίνεται. Η πανικοδόμηση σε εμπορικό, οικονομικό, πολιτιστικό και χρηματιστικό επίπεδο του Ιράκ και να εγγυηθούμε την ασφάλειά του είναι προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, αλλά θα πρέπει να ευνοήσουμε και την ενίσχυση των θεσμών στη χώρα η ειρηνική συμβίωση μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών συνιστοσών και θρησκευτικών πιάτων αποτελεί ε, περνάει μέσα από μια ανακαίνιση των θεσμών και μέσω ομοσπονδιακής λύσης, μέσω ενός φεντεραλιστικού σχεδίου που επιτρέπει μεγάλη αυτονομία των διαφόρων περιοχών ε, στα πλαίσια του κράτους. Το Ιρακινό Κουρδιστάν μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη της ύπατης εκπροσώπου της Βαρόνης Άστον επ' αυτής της θεσμικής πτυχής της χώρας. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κ. Σβένσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε βία και καταστροφές στο Ιράκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι υπάρχει να εξελίξει μια διαδικασία δημοκρατικοποίησης στο Ιράκ. Στις τοπικές εκλογές πέρσι πάνω από 3.000 γυναίκες κατέβηκαν στις εκλογές ως υποψήφοι, κάτι το οποίο είναι μοναδικό για μια αραβική χώρα. Πάρα πολλέ γυναίκε εξελέγησαν σε υψηλά αξιώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια αραβική χώρα. Είναι και μια ελπίση για τις γενικές εκλογές που θα γίνουν στις 7 Μαρτίου του 2010 οι Σουνίτες <clears throat> συμμετέσχαν στις τοπικές εκλογές αλλά πριν από μερικές μέρες 14 Σουνιτικά κόμματα και πάνω από 500 πολιτικοί απαγορεύτηκε η παρουσία τους στις εκλογές. Ο κ. Αρμουτλάκ, ο Υπουργός ε, Άμυνας που ήταν επικεφαλής του Σουνιτικού Κόμματος για το Διαλόγο είναι μεταξύ αυτών των πολιτικών που απαγορεύτηκε να είναι υποψήφοι. Είναι σημαντικό για τη δημοκρατικοποίηση του Ιράκ και για την πρόοδο του Ιράκ να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την εθνοτική και θρησκευτική συνοχή του Ιράκ. Κυρία Αστόν, σας λέω να είμαστε σαφείς εδώ. Όταν μιλάμε για εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες στο Ιράκ, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επάγρυπτοι. Οι εκλογές στο Ιρακινό Κοινοβούλιο είναι αποφασιστικές για το μέλλον του κυρίου Ιράκ. Οπότε κυρία Άστον, η πάτη τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε αυτές οι εκλογές στο Ιράκ να είναι όσο το δυνατόν δημοκρατικές και ελεύθερες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλτσίτης έχει το λόγο για 90 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σημαντικά την επιρροή της στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα έδινε μεγάλη προσοχή στο Ιράκ και μαζί με τη διεθνή κοινότητα συμμετείχε στην ανοικοδόμηση του Ιράκ και την ασφάλεια και την ειρήνη στη χώρα. Βλέπουμε εσωτερικές διαμάχες, πολιτικές διαμάχες στη χώρα που παρεμποδίζουν την πολιτική μεταρρύθμιση σε διάφορους τομείς. Ανησυχούμε επίσης διότι 14 κόμματα απεκλείστησαν από τη συμμετοχή στις εκλογές. Χρειάζεται εκδημοκρατισμός μέσω δημοκρατίας, δημοκρατικών διαδικασιών μάλλον. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα πρέπει να απαιτήσουν τη συμμόρφωση της χώρας ε, με τους διεθνείς κανόνες και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το Ιράκ πιστεύω ότι είναι έτοιμο για στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα στον ενεργειακό τομέα αποδεικνύει ότι το Ιράκ θέλει να αναπτύξει αμοιβαία αποφελή σχέσεις. Είναι πολύ σημαντική χώρα στρατηγικής, από στρατηγικής πλευράς το Ιράκ όσον αφορά τον ασφαλή εφοδιασμό, τον ενεργειακό και σχετίζεται και όμως η κατάσταση στη χώρα με την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΥΠΑ, του, της ΥΠΑ της εκπροσώπου και με τη βοήθεια της διεθνής κοινότητας μπορεί να βρει λύση, ούτως ώστε το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν ο βασικός πολιτικός πυλώνας που στηρίζει το Ιράκ στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαρνέσκη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, <clears throat> κυρία η Πάτη εκπρόσωπος, αντιπρόεδρε της Επιτροπής λοιπόν, κυρία Άστον θα ήθελα να τονίσω ότι τα λόγια σας σήμερα ήταν ένα είδος κρατικής αισιοδοξία, επίσημης αισιοδοξίας αλλά οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν πολύ περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαίω. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο αυτό το οποίο είπατε, υπάρχουν και αυτά τα οποία δεν είπατε και από τα λόγια σας μου λείπει οποιαδήποτε οποιαδήποτε μνήμα του γεγονότος ότι παραπλανείται ένα μεγάλο μέρος της κοινή γνώμη στην Ευρώπη και ακόμα και στη δική μου χώρα. Αναφέρομαι στην καταδίωξη, στην δίωξη των μειονοτήτων στο Ιράκ και ιδίω των χριστιανών στο Ιράκ. Αναφέρθηκε τον κύριο Τορέμπα, ο οποίος έθιξε το θέμα αυτό, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μία παρέμβαση του Ιράν στο Ιράκ. Δεν είναι γεγονός ότι με, σκανδαλο, με σκανδαλώδη τρόπο χρησιμοποιούν οι αρχές του Ιράκ και την παρέμβαση του Ιράν για τους δικούς τους στόχους. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε λοιπόν αυτό, γιατί ο πληθυσμός του Ιράκ και οι Ιρακινές αρχές παίρνουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν χρησιμοποιούνται προς όφελος του πληθυσμού. Grazie. Σας ευχαριστώ. Ξεκινούμε διαδικασία προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου, ΚΑΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Σάνικ έχει το λόγο για ένα λεπτό. <coughs> Μπορεί να, να είναι ένα παράδειγμα το Ιράκ να δείξει πώς μπορεί κανείς να σπάσει τη ραχοκοκαλιά ενός τυράννου. Και νομίζω ότι οι αποφάσεις τέτοιου τύπου είναι δύσκολο να ληφθούν. Βλέποντας τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράκ, να θυμηθούμε κάτι. Ότι χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό είναι τραγωδία και για εκείνους βέβαια και για τις οικογένειές τους. Και νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε ε, έχοντας υπόψη μας το σκοπό που θέλουμε να πετύχουμε και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειές μας για την παγίωση της δημοκρατίας στη χώρα. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η ύπατη εκπρόσωπος και τι μπορεί να πετύχει η Ένωση. Θα πρέπει να επηρεάσουμε τις εξελίξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό οι μειονότητε να προστατεύονται, όπως χριστιανική μειονότητα. Σας ευχαριστώ. και για ένα λεπτό. Ο κύριος και έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που τόσες φωνές συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Δοθέντως ότι είναι σημαντικό το θέμα του Ιράκ και προσπαθούμε να επιβάλλουμε την ειρήνη. Η κατάσταση στη χώρα ίσως βελτιώθηκε κάπως, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ εύθραστη. Και η Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της καταστάσεως. Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η Ένωση, αλλά δεν τα κάνει. Ας δούμε τι γίνεται με την ανάπτυξη και τη σταθερότητα του Ιράκ. Το σημαντικότερο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους νέους Ιρακινούς φοιτητέ που θα μπορούσαν να μάθουν στην, να στην Ευρώπη να μάθουν. Δεν έχουν μηχανικούς, δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν εμπειρογνώμονες στη χώρα. Μπορούσαμε να τους εκπαιδεύσουμε εδώ. Κάτι άλλο πρακτικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε να προστατεύσουμε τις διάφορους, ε, διάφορες πολιτιστικές συνιστώσεις του Ιράκ. Και μπορούμε να κάνουμε κάτι για την ανοικοδόμηση του Βαβυλώνας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζούμπικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το δικό μου το ερώτημα αφορά το κατά πόσον υπογράφει και το μνημόνιο αντίληψη ε, για την ενέργεια. Με τον κύριο ούτε και με τον κύριο Βαντεγκούχτε πιστεύετε ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Θεωρώ ότι η οικονομική ανάκαμψη στο Ιράκ ε, μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα. Και αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις στον ενεργειακό τομέα αφενός ε, με την παράδοση, την προμήθευση περισσότερων μηχανημάτων στο Ιράκ για την καλύτερη χρήση ενέργειας και αφετέρου με την αγορά ενέργειας από το Ιράκ. Αν το κάνουμε αυτό και οι δύο πλευρές ε, θα κερδίσουν και θεωρώ ότι σε αυτό τον τομέα θα έπρεπε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες να αναλυφθούν πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσει, Δίνω εκ νέου το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άστον. Uh, Σας ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αν προσπαθήσω να σταθώ στα θέματα τα οποία έτυχαν του μεγαλύτερου ενδιαφέρον από τα μέλη του Κοινοβουλίου, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία που αποδίδεται στα θέματα των μειονοτήτων. Όπως τα γνωρίζουν τα έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ένα από τα βασικά στοιχεία μας στη συνεργασία με το Ιράκ είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην καρδιά της ενασχόλησής μας. Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει και στη συμφωνία που θα μονογραφήσουμε με το Ιράκ. Αλλά κατανοώ και αναλαμβάνω την ευθύνη να ληφθούν πλήρως υπόψη τα θέματα των μειονοτήτων στο Ιράκ. Εγώ Σημερίζω επίση του στόχου που έθεσαν μια σειρά από αξιότιμα μέλη σε ό,τι αφορά την θανατική ποινή. Ο στόχο μα είναι να καταργηθεί για του λόγου που έχουν πολύ σωστά αναφέρει τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Κατανοώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να εδραιώσουμε το πολιτικό γίγνεσθε στο Ιράκ. Αυτό θα είναι μεγάλη σημασία για το μέλλον και σε όλες τις προσπάθειές μας και να εξασφαλίσουμε ιδιαίτερα ότι στις επερχόμενες εκλογές του Μαρτίου θα υπάρχει πλήρης κατανόηση του τι θέλουμε να επιτύχουμε. Κατανοώ αυτό που είπαν μερικά έντιμα μέλη, ο κύριος Κώστας, ο κύριος Στίβενσον, σε ό,τι αφορά την, εκλογική, την απόφαση εκλογικής επιτροπής που εμπόδισε κάποιους υποψηφίους να είναι παρόντες εκλογές. Βέβαια, υπάρχει πάντα μια τέτοια διαδικασία σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και υπάρχει και μια διαδικασία έφεσης που ελπίζω θα λειτουργήσει σωστά. Εμείς είμαστε έτοιμοι να στείλουμε μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα, έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές, κάτι θα μας επιτρέψει με πρώτο χέρι να παρακολουθήσουμε την προεκλογική διαδικασία η οποία είναι μεγάλη σημασία στο Ιράκ. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι οι Ιρακινές αρχές θα <clears throat> εξασφαλίσουν μια πλήρη και ελεύθερη διαδικασία εκλογών για όλους τους λόγους που έκαναν ιδιαίτερα σαφή, σαφείς τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ορισμένοι βουλευτές έθεσαν το θέμα του μνημονίου κατανόησης για την ενέργεια και τις σημασίες που επέχει αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής η επιχειρηματολογία μας. Το Ιράκ είναι ένα ενιαίο κράτος και όλη η συνεργασία μας θα πρέπει να γίνεται με την κεντρική κυβέρνηση όλων των Ιρακινών. Θέλουμε το Ιράκ να παραμείνει ανεξάρτητο και κυρίαρχο Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει και κατανόηση αυτά που είπαν ορισμένοι όπως ο κύριος Ρούμπιχ ο οποίος ανέφερε την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία με το Ιράκ και <clears throat> θα το μεταφέρω στην αρμόδια επίτροπο ανάπτυξη στο θέμα αυτό. Θέλω να τονίσω όμως ότι υπάρχει και το θέμα αυτό της ασφάλειας. Το θέμα της Κερκούκ είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ιράκ και το μέρος, όπως και η περίπτωση άλλων σύνορων που είναι αμφισβητούμενα. Πιστεύω λοιπόν και είμαι πεπισμένη γι' αυτό ότι το Ιράκ πρέπει να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα για το καλό των Ιρακινών. Αλλά θέλω να τονίσω την απαραίτητη η αρρωγή των Ηνωμένων στο Ιράκ. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες να ξεκινήσει ένας διάλογος και μια διαδικασία στο Ιράκ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν νομίζω ότι πριν από τις εκλογές θα μπορέσει να προχωρήσει ιδιαίτερα ο διάλογος. Κάτι ακόμα θέλω να σας πω σε σχέση με την ενεργειακή συνεργασία με το Ιράκ. Για μας αυτό είναι τμήμα της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ενεργειακής πολιτικής για το Ιράκ. Είναι θέμα παροχής ενεργειακών πόρων και ασφάλειας ενεργειακών πόρων από το Ιράκ στην Ευρώπη και ιδίως ανάπτυξη επίσης ανανεώσιμης ενέργειας που είναι ηλιακή, και αιωλική ενέργεια και μέτρα ε, εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βοηθήσουμε και τη βιομηχανική συνεργασία στο Ιράκ στους επερχόμενους μήνες και τα χρόνια, αλλά κατανοώ αυτό το οποίο είπατε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ακύρωση της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για λόγους ασφαλείας όπως αναφέρθηκε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια βελτίωση στο κλίμα στο Ιράκ ώστε να μπορέσει να πάει η αποστολή παρακολούθηση των εκλογών με τη συμμετοχή βουλευτών, κάτι το οποίο θα είναι πολύ μεγάλη σημασία μέσα στην εκλογική διαδικασία και θα σας δώσουμε στοιχεία γι' αυτό το ταχύτερο δυνατό. Αναφέρθηκε το θέμα της απόσυσης των δυνάμεων από το Ιράκ. Είπε ο κύριος Ομπάμα ότι τον Αύγουστο 2010 δεν θα υπάρχουν μάχημες δυνάμεις στο Ιράκ, οπότε θα αρχίσει η απόσυρση, η αποχώρηση των δυνάμεων σύντομα μετά τις εθνικές εκλογές στο Ιράκ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τόνισα ότι θα στείλουμε μια ομάδα αξιολόγησης των εκλογών στο Ιράκ ως ο Νούπο, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν θέσει τα αξιότιμα μέλη. Και επίσης έχουμε τονίσει στο Ιράκ ότι το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί βάση του διεθνούς δικαίου. Εγώ είμαι πάντως αισιόδοξη σε σχέση με το Ιράκ. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στα έντιμα μέρη του Κοινοβουλίου. Ορθά μας το υπενθυμίζουν, αλλά βλέπουμε ότι με τις επερχόμενες εκλογές, με την ευκαιρία να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, ότι υπάρχει χώρος η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύστημα αξιών τους, με τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των μειονοτήτων, τα θέματα της θανατικής ποινή και όλα αυτά να αναπτύξουμε μια συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και στην παροχή ενέργειας. Ελπίζουμε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα με την κυβέρνηση του Ιράκ, τονίζοντας πάντα ποιε είναι οι προσδοκίες μας ότι θέλουμε ένα Ιράκ το οποίο θα είναι ειρηνικό και δημοκρατικό και θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους προς τον στόχο αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Πέρα στι συζητήσεις Διακόπτεται η σύνοδος μέχρι τις 9 το βράδυ.